Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. S'il vous plaît. συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. La séance Λοιπόν, ξεκινάει η συνεδρίαση. Σήμερα το πρωί έχουμε μια σειρά ψηφοφοριών. Οι δύο πρώτες αφορούν το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, έκθεση πρωτοβουλίας Olbricht Τομά. Η δεύτερη είναι η έκθεση πρωτοβουλίας για τους νέους ίδιους πόρους. Είναι η έκθεση Ντεπρέ και Λεβαντόφσκι. Σας παρακαλώ να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Le scrutin est ouvert. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. 27 ψήφισαν. μάλλον 27 έβαλαν την κάρτα του στο μηχάνημα αλλά δεν ψήφισαν. 26. Ποιος είναι ο 27ος? Αλλά πέρασε. Ωραία. Θα ψηφίσουμε την έκθεση πρωτοβουλίας πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά λοιπόν να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρασε Απορρίπτεται ε, με ευρεία πλειοψηφία. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Και contre. Qui s'abstient κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 13 υπέρ 12 κατά. Α, τελικά απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 129 και 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 131 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτω 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 142 και 143 οι, οι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά Αποχέ, απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 έως 153 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 έχει αποσυρθεί 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100... Να ελέγξουμε. Την 168 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 23 κατά, 11 υπέρ, 169 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 192. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Μέχρι το σημείο άλλα προγράμματα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 228 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα έχουμε τροπολογίες 2.31, 2.30, 2.31, 32, 33, 34 που θα, και 2.35 που θα μπορούσαν να ψηφιστούν μαζί. Αφορούν τις παραγράφους, την υποπαράγραφο 9, την παράγραφο 42 και την παράγραφο 43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 2.36 υπέρ κατά Α, ήταν τμήμα του μπλοκ. Α, μάλιστα. Δεν το είχα αναγγείλει βέβαια, αλλά θα θεωρήσουμε ότι είναι αυτονόητο. 2.37. Ναι, ψηφίζουμε. 2.37 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, 21 κατά. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.65 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 285 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 286 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτε. 3.14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 328 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τριοπολογία 359 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρα. Εγκρίνεται. 19 υπέρ, 15 κατά. 362 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.91 με μια προφορική ε, του, των εισηγητών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4-12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4-13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4-14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 4.15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.16 και 4.17 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 4.18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται συγγνώμη Συμβαστική 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Μάλλον θέλετε λίγη, ένα διάλειμμα γιατί δεν βλέπω να σηκώνει τα χέρια σας. Παρακαλώ. Επομένως 472 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμό 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεθετείτε. Τροπολογία. 496 υπέρ. Κατά. Θα το επαληθέσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 497 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβασμό 46 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 506. Με χωριστή ψηφοφορία το ζήτησαν το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές. Πρώτο τμήμα μέχρι το εξάντε της υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 508 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 510 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 519 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμό 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 530. Σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος μέχρι το Education and Healthcare. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 536 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 535 υπέρ. Όχι καταπίπτει. Συμβασμό 48 υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμό 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία. 556 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 569 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Συμβασμός 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 599 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 612 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 604 υπέρ. Κατά. Θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας προφορίας, Υιοθετείται. 20 υπέρ, 16 κατά. Τροπολογία 628 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 629 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 639 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται 640 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 642 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 644 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζεται τώρα. Την 644. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 22 κατά 14 υπέρ. 645 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 646 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 647 υπέρ κατά θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τώρα πέρας προφορίας 16 υπέρ, 16 κατά. Κύριε Ολμπριχτ, ψηφίσατε. Ναι, ναι. Απορρίπτεται τότε. Στο τσακ. Συμβασμός 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 659 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 660 και 661 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 663 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 662 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 664 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Συμβασμός 56 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 676. Σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα. Μέχρι το gender balance. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το υπερθέψουμε. Ψηφίσουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 22 ψήφικα, τα 14 πέρα. 6,77 σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβασμό 58 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 59 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 591. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Με μια προφορική τροπολογία. Έχετε το κείμενο μπροστά σας, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Υιοθετείτε. 18 ψήφι υπέρ, 16 κατά. Συμβασμός 60. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας καθαρά. Υπέρ ή κατά. Συμβασμός 61 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 62 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Προφορική τροπολογία για την παράγραφο 97 για να προσθέσουμε μια φράση υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 63 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 6,82 υπέρ κατά απορρίπτεται. 6,83 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Η 172 καταπίπτει. 6,78 και αυτή καταπίπτει. Πάμε λοιπόν αιτιολογικές αναφορές. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 8 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 9 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 10 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Αιτιολογική σκέψη τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 64 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 18 υπέρ. Όχι καταπίπτει. Είναι μη παραδεκτή. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Θα την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Την 24. Ψηφίζουμε Πέρες. Πέρες. Ο, απορρίπτεται άνετα. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια. Τροπολογία 25. Καλύπτεται ήδη. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στις αγνομοδοτήσεις της Ρέτζι. Έχουμε διάφορες αγνομοδοτήσεις που καλύπτονται. Ρέτζι C υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αυκό. Δεν πρέπει να ψηφίσουμε. Όλα καλύπτονται. Κοντ. Να ψηφίσουμε συνολικά όλες οι γνωμοδοτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί ήδη. Τις παραγράφους διορθώνε προς που δεν καλύπτονται. Υπέρ. Ο κύριος Ντεπρέ. Θέλετε χωριστή ψηφοφορία. Ωραία, θα ψηφίσουμε χωριστά. Παράγραφος 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Ε, κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα Στι παραγράφου που αφορούν τι αρμοδιότητε τη Επιτροπής Αλίας. Παράγραφος 13 υπέρ. Μπορούμε να τι ψηφίσουμε όλε αυτέ τι παραγράφου που δεν καλύπτονται Όλε μαζί. Κύριε εντεπχέ, τι λέτε. Εκτό από την 29 και την 30. Τις υπόλοιπε μαζί. Ξαναπέστε το με μικρόφωνο παρακαλώ. Πολύ ωραία. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί εκτός από την 29 και την 30. 13 λοιπόν. Από την 13 έως την 27. Ουφ, τώρα με μπερδέψατε. Θα ας ψηφίσουμε μία-μία τις παραγράφους. Παράγραφος 13. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λίμπε α δεν ξέρω την 30 30 υπέρ της πέσα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Λίμπε, όλες καλύπτονται. Τραν, παράγραφος 4, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 12, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 26. Ναι, έτσι πάω γρήγορα γιατί αλλιώ. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Επιτροπή Πολιτισμού, παράγραφος 22 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Επιτροπή Γυναικών, παράγραφος 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε. Παράγραφος 15. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στην αφέτητα έχουμε κάτι. Envy. Παράγραφος 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 επέρ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 επέρ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 επέρ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19 επέρ, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 επέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 Επέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύε από κοινού. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, να ψηφίσουμε την 2, 20, 21, 31, 44, 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και για το σύνολο του εγγράφου, όπως έχει τροποποιηθεί ψηφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. 29 ψηφί υπέρ, 4 κατά. Και 3 αποχές. Εγκρίνονται λοιπόν. Συγχαρητήρια στους δύο συνεισηγητές. Την Ιζαμπέλ και τον Γιάννη. και ευχαριστούμε και τους συνεργάτες και τους κοιόδους συζητητές για την προετοιμασία των συμβαστικών τροπολογιών που σίγουρα ήταν δύσκολη υπόθεση. Ας πάρουμε μια ανάσα. Πίνω λοιπόν λίγο νερό στην υγεία σας. vous invite à boire un coup si vous en ressentez la nécessité.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 Ευχαριστούμε τους δύο συνεισηγητές και τους συνεργάτες τους που προετοίμασαν και τις λίστες ψηφοφορίας και βέβαια τις συμβαστικές. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Τώρα λοιπόν θα ψηφίσουμε την έκθεση της πρωτοβουλίας ε, των Ντεπχέ και Λεβαντόφσκι. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται.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 απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 15, τροπολογία 37. Υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 9, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 16. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σεβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σεβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. σημαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σεβαστική 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. <clears throat> Τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 17 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83 έχει αποσυρθεί. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά Α, ξεχάσαμε την 89. Υπέρ για την 89, κατά, Δεν σηκώνω τα χέρια και δεν καταλαβαίνω. Επομένω, τιμωρία, ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται 20 ψήφοι κατά, 14 υπέρ. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 και 95 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 99 έως και 111 θα μπορούσαμε να τις ψηφίσουμε μαζί, αν θέλετε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 107 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116, 118, 120, 124 126 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 125 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ηλεκτρονικά. Να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 20 κατά 14 υπέρ. Σεβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 27α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 28α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 28β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 28 δέλτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Envy. Amendement 157. Ε, Άμβη 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει 157, συμβαστική 28 ε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά σας παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας άρα θα χρειαστεί ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται επί της 164 ψηφίσατε όλοι πέρασε εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ 14 κατά 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα να περάσουμε στις ιδεολογικές σκέψεις. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στις γνωμοδοτήσεις τη ίντα. Παράγραφοι 5 και 6 δεν καλύπτονται. Θα μπορούσαμε να τις ψηφίσουμε από κοινού. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία. Όπως τροποποιήθηκε το κείμενο, να ψηφιστεί βεβαίως με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Λείπει ένας. Λείπει μία ψήφος. Τελευταία ευκαιρία για τον 36ο να ψηφίσει. Δεν ψηφίσει. Α, ψήφισε. Ευχαριστώ πολύ. Πέρας. Εγκρίνεται 31 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, και μία αποχή. Συγχαίρουμε τον Ζεράρ Πρέ και τον Γιάννους Λεβαντόφσκι, οι οποίοι από κοινού επέτυχαν 31 ψήφους υπέρ. Ωραία. Συγχαρητήρια και στους ε, συνεργάτες μας. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι επειδή ψηφίσατε για το ΠΔΠ και τις νέους ίδιους πόρους, ότι δεν είναι σημαντικές και οι επόμενες εκθέσεις. Τονίζω τη σημασία τους. Λοιπόν, υπάρχει μια τροπολογία... Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον άνθρακα και χάλιβα. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ναι ή όχι. Ονομαστική ψηφοφορία για το κείμενο αυτό που δεν είναι τροποποιήσιμο. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι μου. Πέρας. Εγκρίνεται 28 ψήφοι. Υπέρ, 2 κατά. Και 2 αποχές. Να συγχαρούμε τον εισηγητή. Ναι, ευχαριστώ. Ε, είναι αυτές τις εκθέσεις που δεν τη θέλει κανείς. Σε ευχαριστώ για τα χειροκροτήματά σας. Ωραία.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 Εγκρίνεται 23 ψηφοί υπέρ, 7 κατά. Συγγνώμη, αλλά σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. Τροπολογία 8. Κατά αποχές και πάλι δεν είναι σαφές. Λοιπόν, παρακαλώ, τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Μα είδα περίπου ε, τις ίδιες ψήφους υπέρ και κατά, οπότε ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται. Πέρας. 26 υπέρ και 6 κατά, αλλά εγώ δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Πιείτε λίγο νεράκι. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές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 Α, όχι, το 17 λέει τώρα ο πρόεδρος. Συγγνώμη. 17. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται 14 υπέρ, 18 κατά. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα, το σύνολο του κειμένου, ονομαστική. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 30 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια στο συνάδελφο Μπάιτ. Και τώρα, την έκθεση, μια άλλη έκθεση προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση είναι η έκθεση Εστέβαν Γκονθάλεθ Πόνς για ένα θέμα της Γαλλικίας. Ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τρία. κατά, ε, κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ το έχει στήσει ο συγκεκριτής. κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται για το δεύτερο τμήμα ο ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 15 ψηφί υπέρ 17 κατά τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές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 Το σύνολο του κειμένου τώρα, όπως τροποποιήθηκε, ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Ενεκρίθη 30 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή, συγχαίρουμε τον εισηγητή. Και τώρα, έχουμε το κείμενο του συναδέλφου Ινέζε Βάιντερέι η συμβολή της γεωργίας και ο προϋπολογισμός σε σχέση με τις εταιρικέ σχέσεις. Το σύνολο του κειμένου. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Α, όχι, έχουμε δύο ψηφοφορίες. Η πρώτη αφορά τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται και επί της γνωμοδοτήσεως ονομαστική άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Δύο δεν έχουν ψηφίσει ακόμη. Πέρας. Εγκρίνεται 27 ψήφοι υπέρ. Τρεις ψήφοι κατά. Συγχαίρουμε, την κυρία Βέιντερεϊ. Λοιπόν, τώρα έχουμε τα χρηματοδοτικά μέσα. ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και προοπτικές 2020. Πρόκειται για την δομή των μέσων. Τροπολογία 1 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεν είναι σαφές, άρα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται 22 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 έχει αποσυρθεί. Η 10 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα η 12 είναι προφορική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Ελέγχουμε τη 13. Πέρας. Απο... Απορρίπτεται. 17 ψήφι κατά. 14 υπέρ. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 23 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Για το σύνολο του κειμένου με νομαστική κλίση παρακαλώ. Ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείται με 28 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους κατά. Υπά... Δεν υπάρχουν αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα έχουμε κάποιες μεταφορές. για τον προϋπολογισμό. Τον προϋπολογισμό του 2018. Είναι συνακόλουθες ψηφοφορίες λόγω των δύο θετικών νομοδοτήσεων που εκφράσαμε για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κάποια δικά σχόλια. Ο Γενικός Εισηγητής, όχι Πρόεδρε. Ψηφίζουμε τις δύο πρώτες μεταφορές του προϋπολογισμού του 2018 και όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι η συνέπεια των δύο εκθέσεων που μόλις υιοθετήσαμε, την έκθεση του Esteban González Pons για τους απολυμμένους εργαζόμενους στην περιοχή της Γαλλικίας και την έκθεση του κύριου Πάιτ για τις απολύσεις στη Σουηδία από την Έριξον. Πολύ συγκεκριμένα ήταν για αυτού τους λόγους. Θα ψηφίσουμε πρώτη μεταφορά για τη Σουηδία που προτείνει να μεταφέρουμε 2 εκατομμύρια 130.000 134.000 από το ε, αποθεματικό στην κύρια γραμμή του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης είναι λόγω της έκθεσης που ψηφίσαμε προτείνω να ψηφίσουμε υπέρ και συνεχεία θα ψηφίσουμε τη δεύτερη μεταφορά που προτείνει να μεταφέρουμε 720.000 ευρώ από το αποθεματικό του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση στη βασική γραμμή του προπολογισμού συνέπεια της έγκρισης της έκθεσης Esteban González Pons και αυτό καλύπτει την αίτηση που έκανε οι Ισπανικές Αρχές για τις απολύσεις στην Καλήθεια. Στη Γαλλικία δηλαδή προτείνω να ψηφίσουμε υπέρ τη ε, μεταφορά αυτή. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Γενικό Εισηγητή. Δεν υπάρχουν δικέ παρατηρήσεις. Πολύ ωραία. Θα ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση για την πρώτη μεταφορά. Ηλεκτρονική ψήφος. Ανοίγουμε τώρα την ψηφοφορία. Ψηφίζεται τώρα. Ε, φύγαν διάφοροι βουλευτές, αλλά άφησαν την κάρτα τους μέσα στο μηχάνημα. Ακόμα μια προσπάθεια, παρακαλώ. Πέρας προφορίας. Υιοθετείτε 27 ψήφι υπέρ, 3 κατά. Τώρα, για την δεύτερη μεταφορά, για τη Γαλλικία, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ψηφίζουμε τώρα. Πέρας φοφορίας. Έγκριση. 28 ψήφι υπέρ, 2 ψήφι κατά. Τώρα, πάμε στα άλλα τμήματα. Ο εισηγητής, ο Ρίτσαρντ Ashworth έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο μεταφορές, δύο αιτήσεις μεταφορών η πρώτη αφορά τις τροποποίηση της Επιτροπής των Περιφερειών και το σχέδιο εγκατάστασης. Το δεύτερο μεταφορά ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, για την Επιτροπή των Περιφερειών. Τροποποίηση οργανογράμματος. Ε, από μόνοι μας τους κάνουμε έκτακτους. Ε, εκπροσωπούν αυτό ε, εξοικονομήσεις. 368.000 και 90 cent για 10 μήνες εξοικονομούμε έτσι. Δεν χρειάζεται ψηφοφορία γι' αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι λίγο πιο περίπλοκο γιατί αφορά το... μια μεταφορά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Κοινοβούλιο, η Γενική Διεθνή ΚΟΜ ε, ζήτησε να μεταφερθούν 3 εκατομμύρια ευρώ από τη γραμμή 3242 στη γραμμή 1400 ε, για τη συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις και έχει μεταφερθεί ε, στο, στη γραμματεία και στις πολιτικές ομάδες. Αυτό οφείλεται στις ευρωπαϊκές εκλογές που έχουμε του χρόνου ούτω ώστε να μπορούμε να επιστρέψουμε να προσληφθούν άλλοι 49 ε, υπάλληλοι για θέματα ε, και τα εκλογικά αυτά, την προεκλογική εξατία και την επικοινωνία. Το Νοέμβριο του 2017 το Προεδρείο αποφάσισε να ε, υπάρχει μια αποκεντρωμένη εκστρατεία προεκλογική και γι' αυτό ακριβώς θα γίνουν αυτές τις προσλήψεις. Ε, πρέπει να ψηφίσουμε γι' αυτό. Ξέρω ότι διάφοροι από εσά είχατε διάφορες ανησυχίες και εγώ το ίδιο και στείλαμε μια επιστολή στη Γενική Διεύθυνση που, την αρμόδια και ζητήσαμε κάποιες διευκρινήσεις. Μοιράσαμε την απάντηση της ε, Digicom που είναι ικανοποιητική. Απάντηση στα ερωτήματα που είχαμε. Το απογοητευτικό είναι ότι εμείς ως ε, οργάνωση χθες συζητήσαμε την προεκλογική εξαρτία το 2019 στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2018. Το Προεδρείο έχει αποφασίσει αυτή την αποκεντρωμένη εκστρατεία. Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό. Ε, μίλησα με τον Πολ Ρούμπικ και νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Οι συνάδελφοι Έλαβαν τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθεσαν όμως, παρόλα αυτά. Χρειάζεται να ψηφίσουμε γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει, δεν θα πρέπει κάτι την απόψή μου να είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη μεταφορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντότζ Γκυγιό είναι παρόν στην αίθουσα, που είναι Γενικός Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ. Πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο να μιλήσει για να καλμάρει τα πνεύματα. Το γεγονός ότι ψηφίζουν δηλαδή έναν προπολογισμό και πριν το τέλος καν του προϋπολογισμού του 2007, ε, στην πραγματικότητα ζητάμε μια τροποποίηση αυτού του προϋπολογισμού, πριν ολοκληρωθεί δηλαδή αυτή, αυτός ο προϋπολογισμός. Τα περισσότερα ερωτήματα έχουν απαντηθεί ε, βασικά έχουμε στείλει μια επιστολή στην Digicom και λάβαμε ικανοποιητικέ απαντήσεις. Διάφοροι συνάδελφοι είχαν επιφυλάξεις. Μπορεί να ήθελαν κάποιες διευκρινήσεις. Και αν η Γενική Διεύθυνση COM, α, μια και είναι εδώ, μπορεί να θέλει να μιλήσει κιόλας για αυτό το θέμα. Υπάρχουν ερωτήσεις. Δεν βλέπω. Πρόκειται για, για τη μεταφορά αυτού του ποσού. και πρέπει να την ψηφίσουμε αυτή τη μεταφορά. Για τις 49 θέσεις αυτές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Υπάρχει μια κάρτα η οποία δεν ξέρω ποιος την έχει. Ε, περνάει με 23 ψήφους υπέρ, 5 ψήφου κατά. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Επιτροπής των Περιφερειών, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα θεωρήσω ότι η Επιτροπή μας υιοθετεί, εγκρίνει αυτή την πρόταση. Σε ό,τι αφορά την πολιτική και τα κτίρια, δεν ψηφίζουμε. Και κατά συνέπεια, τελειώσαμε τη για διάταξη. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 8 Μαρτίου από τις 9 μέχρι τις 12.30. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που ήρθατε όλοι εδώ σήμερα το πρωί για αυτές τις σημαντικές ψηφοφορίες που έχουν να κάνουν με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.